του δικαίου, διάρκεια μία ώρα το όριο, άρθρο 122 του κανονισμού. Πρώτο θέμα στα κατεπήγοντα κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Έχουμε ψηφίσματα και θα μιλήσουν πρώτα οι συντάκτες με πρώτο τον κύριο Ρωμέβα Ιρουέντα. Thank you so much, ε, Σας ευχαριστώ. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ανησυχούμε για την κατάσταση στην Αφρικανική Δημοκρατία που είναι σε κατάσταση έκρηξης με σημαντικές επιπτώσεις στο πληθυσμό από τότε που η Σελέκα πήρε το Μάρτιο την εξουσία η αυξημένη βία μεταξύ των κοινοτήτων και θρησκευτικών ε, πίστεων έχουν οδηγήσει σε μία έκρηξη της πολιτικής κατάστασης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαιλασία, σεξουαλική βία κατά των γυναικών, αυθαίρετα της φυλακίσεις ε, και στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών ε, παρά τις προσπάθειες να ε, αντιμετωπιστεί ο πόλεμος μεταξύ των θρησκειών και μεταξύ των κοινοτήτων θεωρείται ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση, εκτός και να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Εμείς λόγω όλων αυτών αλλά και πολλές άλλες ομάδες έχουμε ζητήσει από τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσουν τις διεθρωτικές αιτίε της σημερινής κρίσης και να συνεργαστούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας της Λιμπρεβίλ προκειμένου να υπάρξει ειρήνη και δημοκρατική λύση μακροπρόθεσμα. Καλωσορίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, ε, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την προστασία των πολιτών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μέσω της στρατιωτική γαλλικής Αποστολή ε, και καλούμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο ε, και καλούμε να έχουν όλοι οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ελεύθερη πρόσβαση σε Όλους όσους υποφέρουν επίσης ε, καλούμε για διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ε, του διεθνούς δικαίου που έχει παραβιαστεί στη χώρα και ζητάμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το εμπάργκο των όπλων για την και Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέβα Ιρουέντα. Και τώρα ο κύριος Μπίλαν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ε, σε επεισόδια στον Μπαγκούι. Επίσης ε, ε, έχουν χάσει τη ζωή τους από άγνωστους ε, σκοπευτές ε, και κάποιοι αλλοδαποί. Η Σελέκα, τη μουσουλμανική αυτή ομάδα, προβαίνει και σε κατά του χριστιανικού πληθυσμού κατάσταση γίνεται όλο και πιο δεινή και η περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης θα οδηγήσει σε μαζικές δολοφονίες λόγω θρησκείας και πρέπει να ε, καταγγείλουμε αυτή τη βία, να ξεκινήσει διάλογος, οι δράστες ε, να ε, τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη και πρέπει να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό χρειάζεται οι διεθνείς οργανώσεις να κινητοποιηθούν. Βασίζομαι λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη για να προστατεύσουν, να εξασφαλίσουν τις βασικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού. Ευχαριστώ η κυρία Ντέκεζερη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να αποτέσω φοροτιμή στου δύο Γάλλου στρατιώτε οι οποίοι έχασαν τη ζωή του στην Κεντρική Αφρική. Και να σα πω ότι σήμερα πραγματικά θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για το ότι μετά από πάνω από ένα χρόνο προειδοποιήσει ε, και προ την κυρία Γεωργίευα και προ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράση χρειάστηκε τόσο χρόνο ε, ώστε να υπάρξει ψήφισμα του ΟΗΕ για να γίνει επιτέλους κάτι, να προστατευτεί η κεντροαφρικανική δημοκρατία. Το ξέραμε, το ξέραμε και το ξέρουμε ότι υπήρχε απειλή για πραγματική γενοκτονία με όλες αυτές τις βιοπραγίες και τις ομότητες ε, που βλέπουμε και έχουμε δει και κατά το παρελθόν. Το γνωρίζαμε αλλά χρειάστηκε πολλής χρόνος για να γίνει κάτι σήμερα. Άκουσα πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για τη δική μου πολιτική ομάδα, να γίνεται λόγος για το ότι ε, αναγεννάται η σχέση Γαλλίας-Αφρικής ε, Γαλλική Αφρική σε σχέση με τη γαλλική δράση και τα λοιπά. Αλλά πραγματικά ε, ουσιαστικά νομίζω ότι η Γαλλία αυτή τη φορά απλά άκουσε αυτά που τόσο καιρό λέμε ορισμένοι από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντεκεζέ. Ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι η τρίτη φορά που συζητάμε την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία φέτος και ε, αυτό για να τη δράσουμε στην αδυναμική της βίας ε, και στα αντίπεινα, τα θρησκευτικά που λαμβάνουν τώρα χώρα. Εγώ επίσης ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Γαλλία είναι εκεί, όχι η Ευρώπη. Η Ευρώπη παρόλα αυτά έχει δείξει την υποστήριξη τις τελευταίες μέρες γιατί επεμπλοκάραμε 500.000 ευρώ για την αποστολή αφίσμα και η Ένωση υποστήριξε επίσης τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής ενέργειας γέφυρας ε, μέχρι τον Μπάνγκη. Η κυρία Ντεκέισερ υπογράμισε ότι η Επίτροπος Γεωργίευα επεσήμανε το ζήτημα, έχει επισημάνει το ζήτημα εδώ και καιρό και τώρα θα πρέπει να αναλάβει δράση γιατί οδηγούμαστε προς μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, πολύ πιο σοβαρή από αυτή που φαντιζόμαστε την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ και με διόρθωση 50.000 το ποσό. Ευχαριστώ η κυρία Βεζιά, για δύο λεπτά. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι από τότε που μπήκε το ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη ε, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στην κοινωνική δημοκρατία. Τρίτη φορά το συζητάμε. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, που πέρασε από τη μία δικτατορία στην άλλη, δεν έχει συγκινήσει του βουλευτέ. Και η δικτατορία αυτή ε, δημιουργήθηκε και με, εγκαταστάθηκε με την αισιοπηρή συνενοχή τη ε, γαλλική ε, κυβέρνηση. Μία από τι ενέργειε στρατιωτικέ βάσει αποτελούν τη βάση για μία από τι τις ε, ε, εκατοντάδες επεμβάσεις της γαλλικής κυβέρνησης. Και εδώ και εβδομάδες προετοιμάζονταν οι γαλλικές δυνάμεις να επέμβουν και τελικά αυτό ε, όξινε και τα πράγματα στο Μπανγκί. Δηλώνουν ότι θέλουν να καταπολεμήσουν τις δράσεις της Σελέκα. Έχουν σπείρει το θάνατο στο πέρασμά τους και ξεκίνησαν ένα σπιράλ βίας. Είχαμε μέσα σε λίγη λίγες ώρες εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, κατοίκους ε, νεκρούς. όμως τώρα έχουμε τον πληθυσμό που έχει δικαίωμα στην ασφάλεια και ναι, έχουμε Γάλλους στρατιώτες που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους, όμως το ψήφισμα θα θέλαμε να μιλάει για το μέλλον, για το μέλλον των πολιτών της Κεντροαφρικανής Δημοκρατίας που τελικά θα έπρεπε και αυτοί να έχουν ένα δικαίωμα να ακουστεί η φωνή τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βεζιά. Θα είχατε 20 δευτερόλεπτα ακόμα, μιλούσατε λίγο πιο αργά για να καταλάβω κι εγώ λίγο περισσότερο αυτά που λέτε πέμπτη απόγευμα. Επιτρέπετε ερώτηση από τον συνάδελφο Πρέντα με την γαλάζια κάρτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βερζιά, κατανοώ ότι διαφωνείτε με την επέμβαση. Η δικιά σας εναλλακτική πρόταση όμως ποια είναι. Αν είναι κακή επέμβαση, εσείς πολύ συγκεκριμένα τι θα προτείνατε να γίνει. Εσείς ίδια τι θα κάνατε ε, σε αντίστοιχη περίπτωση. Κύριε Πρέντα, συνήθως με ακούτε προσεκτικά. Ποτέ δεν απεφάνθηκαν κατά της στρατιωτικής επέμβασης. Λυπούμε που αναγκαζόμαστε να επεμβαίνουμε με τέτοιο τρόπο. Και ακριβώς απέναντι στη διεθνή ε, απάθεια είναι εύκολο να πει κανείς θα επέμβει Γαλλία. Εδώ και ένα χρόνο ζητήθηκε ψήφισμα από τον ΟΗΕ δεν είναι ικανοποιητικά. Η πρώην Αφρικανική δύναμη που δεν έχει ακόμα συσταθεί του ΟΗΕ τόπου δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι ε, διεθνής η αδράνεια και συλλογική ευθύνη. Δεν είπα τίποτα για τη στρατιωτική επέμβαση. Απλώς είπα ότι λυπούμε γιατί έχασαν τη ζωή τους δύο Γάλλοι στρατιώτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερζιά. Η κυρία Γιάτεμάκη. Arvoisa puhemies, Kuten Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως έγινε η γαλλική αυτή επέμβαση, όχι η ευρωπαϊκή, είναι σε εξέλιξη. Ε, γαλλική επέμβαση, ο Φρασουά Ολάντα δήλωσε ότι είναι μεν επικίνδυνη αλλά απαραίτητη αυτή η επέμβαση. Όπως όλοι και εγώ ανησυχώ με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Τα πάντα λείπουν και η τροφή και κυρίως βέβαια η ασφάλεια. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία βλέπει να πηγαίνουν σχολείο πολύ λίγα παιδιά. Ούτε ε, μπορούν να τραφούν σωστά τα παιδιά. Τα πιο πολλά υποσυτίζονται. Έχουμε ανθρωπιστική ε, δυσκολία. Έχουμε μάλλον πρόβλημα ανθρωπιστικό, χρειάζεται βοήθεια. Αλλά η βοήθεια πρέπει να φτάσει εκεί που πρέπει. Χρειάζονται επίσης και πολιτικές παρεμβάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την εξέβρεση ειρηνική λύση. Ευχαριστώ. Μέχρι εδώ ήταν οι συντάκτες. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Σόνικ, για ένα λεπτό. Η σύραξη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κλιμακώνεται. Ε, στρατό τη ε, Σελέκα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσφεύγει σε βιοπραγίες. Τα θύματα αυτών των βιοπραγιών είναι συνήθως γυναίκες και παιδιά. Στις 5 Δεκεμβρίου για 72, σε 72 ώρες 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και είναι πιο ανησυχητικό ότι τέτοιες ε, βιοπραγίες διαπράττονται από εγκληματικέ ομάδες ε, που είναι ε, βαριά οπλισμένες και καλωσορίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη σκοπεύουν να στείλουν μια ειρηνευτική αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε επίση να συμμετάσχει στις προετοιμασίε για μια πολιτική λύση, για ένα πολιτικό σχέδιο για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προκειμένου να υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόνικ. Ο κύριο Δεζίρ για 1,5 λεπτό. Merci, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από τότε ε, που η ΣΕΛΕ την εξουσία στις 24 Μαρτίου 2013 ε, οι βεοπραγίες ε, έχουν, βασ... έχουν βυθίσει την κεντροαφρικανική δημοκρατία σε ένα σπιράλ βίας. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει την αιστεία τους και είναι δραματική ανθρωπιστική κατάσταση. Ήταν λοιπόν επίγον να αναλάβουμε δράση και αυτή την απόφαση έλαβε ομόφωνα το Συμβουλίο Ασφαλείας και σε βάση τη εντολή των ΗΠΑ παρεμβαίνει η Γαλλία δίπλα στις αφρικανικές δυνάμεις με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν και στηρίζουν τη Μίσκα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τις πολιτοφυλακές. Εγώ χαιρετίζω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ τη Γαλλική επέμβασης και εγώ αποτείω φοροτιμή στους δύο Γάλλους στρατιώτε ε, που έχασαν τη ζωή τους ε, εδώ από σήμερα. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη και καθολική απάντηση που να απαντήσει και στις απαιτήσει της ασφάλειας, στην ανάπτυξη, στην πολιτική μετάβαση και την οργάνωση ελευθερών εκλογών. Σήμερα χρειαζόμαστε την πλήρη ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά τα επίπεδα για να απαντήσει στην κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω να ακουστεί. Ευχαριστώ κύριε Δεζέ. Ο συνάδελφος Τάκουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι πραγματικά δύσκολη και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να στηρίξουμε την ειρηνική ανάπτυξη την ειρήνευση ουσιαστικά, την, τον τερματισμό της βίας. Μια βία πολύ ομή, ιδίω κατά παιδιών. Υπάρχουν επίσης εγκλήματα πολέμου που βλέπουν να διαπράττονται. Πρέπει κάπω να βοηθήσουμε και εμεί να επανέλθει, να αποκατασταθεί η ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί μαζί και με την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό μέσο να ενισχυθεί και η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή αυτή για να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση με τον τρόπο αυτό και βέβαια να βοηθήσουμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό οι διαφορετικές θρησκευτικέ κοινότητες ε, να ε, συζητούν μεταξύ τους, γιατί μόνο με αυτό το διάλογο θα πετύχουμε και σταθεροποίηση και ειρήνευση στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Σπάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επί

ένα έτος τώρα στην ε, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία διάφορες πολιτοφυλακές συγκρούονται μεταξύ τους και τρομοκρατούν ε, τον άμαχο πληθυσμό. Οι αρχές της χώρας δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των αμάχων. Ακόμα και οι αφρικανικές δυνάμεις ε, που αναπτύχθηκαν εκεί δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν την τάξη. Γι' αυτό ο μόνος κατάλληλος τρόπος προστασίας της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών είναι η εφαρμογή του ε, ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ και ενίσχυση της διεθνούς αποστολής ε, με ανθρωπιστική βοήθεια ενισχυμένη επίσης έτσι ώστε μαζί με την αποκατάσταση της τάξης στη χώρα να έχουμε και αρκετά τρόφιμα για το λαό. Είναι φτωχοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέτσου για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από λιγορή 8 μηνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα που θα αποτρέψει την καταστροφή της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ως κράτος. Ε, εκεί ε, υποφέρουν από λοιμό 1.300.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 300.000 είναι πρόσφυγες. Θα πρέπει το συντομότερο να στέλνουμε ε, τρόφιμα εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να φροντίσει για την προστασία του ομάχου πληθυσμού. Έτσι ώστε ε, να έχουμε αποτελέσματα. Για να έχουμε αποτελέσματα όμως θα πρέπει να είναι ειρηνευτικές οι δυνάμεις ε, εκεί, ε, οι στρατιωτικές, αλλά να υπάρχει και ένας πολιτικός βραχίωνας για να προωθηθούν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Οι ατέρμονες συγκρούσεις στη χώρα αυτή την έχουν διαλύσει, την έχουν διχάσει και επίκειται θρησκευτικός πόλεμος. Ευχαριστώ κυρία Κρέτσου. Ερχόμαστε στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα να δώσω λόγο σε όλους τους συναδέλφους που το ζήτησαν. Η κυρία Χίμπνερ. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι κλασικό παράδειγμα μιας χώρας που παρά τις οικονομικές δυναμικές της έχει εμπλακεί σε θρησκευτικέ και πολιτικές σειράξεις και έχει γίνει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Υποφέρει από οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχουν ολοένα και μεγαλύτερες συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμανών και χριστιανών. Υπάρχουν βασανιστήρια, σεξουαλική βία, εκτελέσεις πολλοί διεθνείς οργανισμοί και τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και πολύ καιρό προειδοποιούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η κατάσταση σε ανοιχτό θρησκευτικό πόλεμο και μαζικές δολοφονίες. Όλες οι προσπάθειες να ανακουφιστεί η κατάσταση δεν εστέφθησαν με επιτυχία. Και βρισκόμαστε τώρα σε κατάσταση ότι χωρίς εξωτερική παρέμβαση θα καταστεί ακόμη πιο βιαφτιά η κρίση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Χίπνερ. Η κυρία Στάιλερ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κλιμακούμενη κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εξακολουθεί να μας ανησυχεί. Και όχι μόνο εμάς και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της μετά από τις διαδηλώσεις αυτές των ανταρτών σε ΛΕΚΑ ε, έχουμε καθημερινά τέτοια πεσόδια βίας, ε, τις 400 τελευταίες δολοφονίες ε, έχουμε βέβαια και μάχες των των που είναι μουσουλμάνοι με τους χριστιανούς υπάρχει μια θρησκευτική βία η οποία οδηγεί σε αποσταθεροποίηση και μπορεί να κινδυνεύει η περιοχή αυτή και με γενοκτονία 50 εκατομμύρια ευρώ βοήθειας, 1.600 ε, ε, Γάλλοι στρατιώτες ε, μετά από ψήφισμα του ΟΗΕ, αλλά η παρουσία της, των δυνάμεων ασφαλείας δεν έχει συγκρατήσει την κρίση και χρειάζεται άμεση δράση για την αποκατάσταση της ειρήνης, της ένομης τάξης. Και η Διεθνής Αμνηστία έχει πει ότι είναι πραγματικά ανευπροηγουμένου κλίμακα των βιοπραγιών και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει επίλυση και ειρήνευση και να λυθεί αυτή η τεράστια κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στάιλερ. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο τώρα, τον κύριο Τσόλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρετίζουμε την παρακολούθηση του Κοινοβουλίου για την κατάσταση και Κεντροαφρικανική Αφρικανική Δημοκρατία και την εθέτηση ενό ψηφίσματο σε σχέση με τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου, τη κατάσταση του κράτου δικαίου. Η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που περνά τη χειρότερη κρίση στην ιστορία τη είναι πραγματικά κάτι ενισχυτικό επανειλημμένα και την τελευταία φορά στις 5 Δεκεμβρίου η ΠΑΤΕΚ πρόσωπος ε, εξέφρασε έντονες ανησυχίες σε σχέση με την κλιμάκωση της βίας ε, και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται με πάσα τιμωρησία. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράζονται στο δικό σας ψήφισμα και ε, αντί της σοβαρότητας κατάστασης πρέπει η διεθνή κοινότητα να δράσει γρήγορα για να αποφύγουμε να εκφυλιστεί κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να επιφέρει μία απάντηση σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο ασφάλειας και ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να συνεισφέρει στην επίλυση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διευκόλυνση του διεθνού συντονισμού μεταξύ των κυριων εταίρων των Ηνωμένων Εθνών της Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΥΠΑ, τη Γαλλία, την Οικονομική Ένωση των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής, η αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και η προστασία του πληθυσμού μένει πολιτική προτεραιότητα. Χαιρετίζουμε την επέμβαση ε, της Αφρικανικής Ένωσης που στηρίζεται από τη Γαλλία και απο ολα άλλα κράτη-μέλη για να τεθεί τέλος ε, στη βία και να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει δεσμευτεί να ενεργοποιήσει, όπως αναφέρατε, 50 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ε, μέσου για την Αφρική για τη Μίσκα. Χαιρετίζω επίσης την υιοθέτηση του ψηφίσματος 2127 από το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΙΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, εργάζεται υπέρ μια στενής παρακολούθησης των εξελίξεων στην ε, Κεντροφυκανική Δημοκρατία μέσω του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενέβη. Η υποστήριξη είναι μορφή Επίσης, ε, συμπεριλαμβάνεται μία επίγουσα βοήθεια προς τους άπορους οι οποίοι αυξάνονται και δράσεις μεσοπρόθεσμες καθώς και ένα έκτακτο μέτρο βοήθεια υιοθετήθηκε από την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος σταθεροποίηση μέσω του μέσου σταθερότητας αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι διάφορες συνιστώσεις στοχεύουν στο να ευνοήσουν την εθνική συμφιλίωση και τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών, μεταξύ των κοινοτήτων, ε, να ε, αναπτυχθούν κάποιοι παρατηρητέ ε, με τη συνεργασία της ΥΠΑ των Ηνωμένων Εθνών και να αποκατασταθούν ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση για να έχουμε αντικειμενική πρόσβαση στην ενημέρωση. Η Κομισιόν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Δράση, επίση εργάζεται μια προσέγγιση Relief Rehabilitation and Development για να αποκαταστήσει τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά μέσα επιβίωσης στη χώρα αυτή. Εξάλλου, η συνεργασία μας για την ανάπτυξη δεν έχει ποτέ αναστολή, ακόμη και αν για λόγους ασφαλείας ορισμένα προγράμματα έπρεπε ε, να παγώσουν. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα θέλει να παρακολουθήσει την διαδικασία μετάβασης. Ε, θα είναι μακρά η διαδικασία αυτή και θα χρειαστούν κοινέ προσπάθειες. Δεδομένες τη πολυπλοκότητα και του εύρου των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, θα είναι καθοριστικό η διεθνή κοινότητα να διατηρήσει τι δεσμεύσει τη εις βάθο χρόνου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίση την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 16 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παραμένει ενεργή για να υποστηρίσει στενό συντονισμό με τους εταίρους σταθεροποίηση της Κεντροαφρικανική Δημοκρατίας και βιώσιμη έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόλο. Έξι συνολικά ψηφίσματα έχουν υποβληθεί προ ολοκλήρωση τη συζήτηση αυτή. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και μετά το τέλος των συζητήσεων θα γίνει ψηφοφορία. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάρκεια.